Just because Good morning everybody. So... Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις ε, πρόεδρων. Πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της 21ης Οκτωβρίου. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, εγκρίνονται. Και περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Και ψηφίζουμε το κείμενο που συμφωνήθηκε στον τριμερή διάλογο για την ταξινόμηση. Δοκιμαστική ψηφοφορία πρώτα. Ψηφίστε παρακαλώ δοκιμαστικά για να δούμε αν δουλεύει καλά το μηχάνημα. Πέρα τη ψηφοφορίας. Ωραία, νομίζω ότι η δοκιμή πήγε καλά. Οπότε Τώρα θα ψηφίσουμε στην πραγματικότητα για τον τριμερή διάλογο. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις 5 85 υπέρ 16 κατά. Εγκρίθηκε και 5 εποχές. Εγκρίθηκε. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.